Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Η συνεδρίαση μας θα διαρκέσει μία ώρα και θα εξετάσουμε το έγγραφο εργασίας από τους δύο συνεισηγητές μας, τον ε, Κόφοντ και τον Γέτσεκ. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες και υποβλήθηκε νομίζω το Δεκέμβριο και νομίζω ότι κατά τη συνεδρίασή μας την Τρίτη με, τις, ε, με τους δύο κύκλους ομιλητές, ομιλητών ήταν ιδιαίτερα ε, χρήσιμες, ε, ιδίως ε, κατά την πρώτη συζήτηση προέκυψαν νέα στοιχεία που πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω. Χθε ε, έγινε συζήτηση στην ΕΚΟΝ με τον Υπουργό Οικονομικών της Μάλτας, ακόμη και εκεί στο τέλος της συζήτησης και της κατόπιν συζητήσεις κατέστη σαφής η διαθεσιμότητα της κυβέρνησης της Μάλτας να συνεργαστεί μαζί μας για να υπάρξει ένα πολύ καλό πρόγραμμα για την προετοιμασία της επίσκεψής μας που θα έχει μεγάλη σημασία. Όμως ε, η συνάντηση της ε, δικής μας Επιτροπής μαζί με την ΕΚΟΝ για να συζητήσουμε με την ε, Μαλτέζικη και την επικείμενη Εστονική Προεδρία δεν κατέστημα λοιπόν δυνατόν να γίνει λόγω μιας απόφασης του Συμβουλίου μια απόφαση του Κορεπέρ ότι το επίσημο πρόγραμμα ε, της Μαλτέζικης Προεδρίας θα παρουσιαστεί αργότερα στην ΕΚΟΝ. Γι' αυτό χρειάστηκε να αναβάλουμε. Αυτό όμως δεν είναι δείγμα καλής συνεργασίας. Μάλλον να ματαιώσουμε. Νομίζω ότι όμως παρόλα αυτά η συνεργασία μας με την ε, Μαλτέζικη Προεδρία είναι σε καλό δρόμο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε αυτό το workshop ε, για τις υπεράκτες δραστηριότητες και την ε, νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος. Τελευταίες εξελίξεις. Ε, η συνεδρίαση αυτή θα γίνει 2 με 4 και θα προεδρεύσουν οι δύο συνεισηγητές. Ε, λοιπόν, εάν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο, να δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές μας. Παρακαλώ, ο Τζέπε Κόφορτ και ο Πίτερ Γέτσεκ. Ποιος θα πάρει πρώτο το λόγο, ο Ζέφερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Συγγνώμη. Είναι σημαντική η συνάντηση για να θέσουμε ε, το ζήτημα της διαφάνειας ε, ε, εκ μέρους των συνεισηγητών για το τι κάνουμε. Γνωρίζετε ότι πρόκειται για μια εξεταστική επιτροπή και είναι ζωτική σημασία να υπάρχει συνεργασία και να συλλέξουμε τα στοιχεία των εγγράφων του Παναμά και να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε στην καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και οι προσπάθειές της για τη δημιουργία διαφάνειας. Ε, σκοπός του εγγράφου είναι να περιγράψουμε το έργο της Επιτροπής μέχρι στιγμής και να καθορίσουμε τις ε, προτεραιότητες μας ως συνεισηγητών. Γι' αυτό ε, συγκαλέσαμε και ε, συνάντηση σκιωδών πριν από τα Χριστούγεννα προκειμένου να υποβάλλετε και εσείς προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το έγγραφο αυτό. Σας ευχαριστούμε για όλα τα σχόλια που λάβαμε. Προσπαθήσαμε ε, να τα ε, εντάξουμε στο έγγραφο που έχετε πλέον. Σας καλέσαμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτών των εργασιών και στη σημερινή συνεδρίαση. Θέλουμε σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας το έγγραφο εργασίας αυτό. Ε, το έγγραφο αυτό προκύπτει βεβαίως από την εντολή της Επιτροπής μας. Έχουμε χρησιμοποιήσει πληροφορίες που συλλέξαμε μέσω των ακροάσεων που έχει διοργανώσει η Επιτροπή μας. Ε, υπήρξε ένας μακρύς κατάλογος ε, εξαιρετικά χρήσιμων ε, ακροάσεων για τα Panama Papers με δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες. Ε, υπήρξε και μια δημόσια ακρόαση για τα διεθνή πρότυπα όπου συμμετείχαν και διακυβερνητικοί διακρατικοί ε, οργανισμοί, ο ΣΑ, ο ΙΕ ε, ε, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων με την ε, Επίτροπο Γιούροβα, ακροάσεις για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Προσκαλέσαμε τον κύριο Μοσκοβισή, τον κύριο Στίγκλιτς, για να μας ενημερώσουν σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτά τα ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, ανταλλαγή απόψεων με τον Άχη Σκούμα ε, που, ε, της FATF, ε, της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Δράσης. Έχουμε κάνει πολλά. Θα συνεχίσουμε με ακροάσεις για τους ενδιάμεσους, καθώς και με αποστολές στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα. Πολλές ακροάσεις Πολλέ ε, πληροφορίε από τι ε, πληροφορίε που λάβαμε βεβαίω ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στο έγγραφο εργασία. θα το κάνουμε όμω εν καιρό. Υπάρχουν έξι κεφάλαια, δεν θέλω να σα τα παρουσιάσω με λεπτομέρειες γιατί φαντάζομαι ότι τα έχετε διαβάσει προσεκτικά. Θέλω όμω να τονίσω κάποια ζητήματα που σχετίζονται με αυτό το έγγραφο. Πρώτον, για μας είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι έχουμε δει ότι οι ενδιάμεσοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σκάνδαλο των ε, εγγράφων του Παναμά και γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς. Το ίδιο ισχύει ε, για το έλλειμμα διαφάνειας καθώς και το ζήτημα της ε, πραγματικής κυριότητας των πραγματικών δικαιούχων ε, το οποίο και έχουμε διερευνήσει όπως θυμάστε στις ακροάσεις μας. Επίσης, θέλουμε, θέλω να ε, εξετάσουμε το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων και των παραδείσων απορρίτου. Το είπε και ο Τζόζεφ Στίγκλιτς ε, η φορολογική παράδεση, η παράδεση απορρίτου είναι η μαύρη πλευρά της παγκοσμιοποίησης και πρέπει να γίνουν ενέργειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Και βεβαίως διεθνής ε, διάσταση, η Μονσέκα Φως δεν είναι βεβαίως η μοναδική εταιρεία που έκανε τέτοια πράγματα, πρόκειται για την κορυφή του παγόβουνου και μόνο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια παγκόσμια οπτική για το ζήτημα αυτό. Αυτά λοιπόν ε, τονίζουμε μεταξύ άλλων στο έγγραφο εργασία μας. Θέλω επίσης να πω ε, εισαγωγικά ότι γνωρίζουμε ότι ε, το έγγραφο αυτό είναι, και το έργο συνολικά είναι πάρα πολύ φιλόδοξο της διερεύνησης των καταγγελωμένων παραβιάσεων. Είναι δύσκολο. Παρόλα αυτά, όμως, έχουμε αποδείξει εδώ στο Κοινοβούλιο ότι ε, θεωρούμε πολύ σημαντική την υπόθεση αυτή και έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο για την ε, διερεύνηση και ελπίζω, είμαι βέβαιος μάλλον, ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο και χρήσιμο ε, κείμενο. Επομένως αξίζει να αφιερώσουμε τον χρόνο και τις προσπάθειες προκειμένου να φωτίσουμε ε, όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα έγγραφα του Παναμά, την ε, φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ε, που θα μας χρησιμεύσει και στο περαιτέρω έργο μας στις άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Αυτά. Από μένα, Πέτρ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πίτερ Γιάτσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σχολιάσω αυτά που προείπατε σε σχέση με την ακύρωση της συνάντησης με τους Μαλτέζους. Χτες όμως, όταν ο Υπουργός Οικονομικών της Μάλτας παρουσίασε τις προτεραιότητες στην Ίκον, πολλοί έθιξαν το ζήτημα της νομιμοποίησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Άρα δεν ξέφυγε δεν μας ξέφυγε. Εν πάση περιπτώσει όμως θα συνεχίσουμε τις ανταλλαγές με την Προεδρία. Ως προς το έγγραφο εργασίας, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά συναντήσεων, ε, επιτόπιες ε, έρευνες και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και θέσαμε το ζήτημα του κατά πόσο πρέπει να έχουμε ένα έγγραφο εργασίας τώρα. Το υποβάλαμε στους σκιώδεις και εντάξαμε όλα τα σχόλια στο κείμενο. Όπως βλέπετε, το έγγραφο σχετίζεται με γεγονότα σε σχέση με τα έγγραφα του Παναμά και είναι ένας οδικός χάρτης κατά τα υπόλοιπα που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε για να φτάσουμε στους στόχους της Εξεταστικής Επιτροπής. Έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πώς ε, δηλαδή ενισχύεται και τι συνέχεια δίνεται από τα κράτη-μέλη και βεβαίως ε, οι διώξεις που γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Σε σχέση με τους ενδιάμεσους είδαμε ότι ε, είναι, βρίσκονται στο επίκεντρο του συστήματος και σχετίζεται βεβαίως με το θέμα της πραγματικής ιδιοκτησίας, νομιμοποίησης χρήματος και ανταλλαγής πληροφοριών. Υπάρχει και η διεθνής διάσταση και τη μελλοντική ερευνητική διαδικασία. όταν ε, πρόκειται για ειδικέ ε, επιτροπές. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης και τη Γραμματεία για τη συνεργασία τους. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε τους Σκιώδης. Ο κύριος Νίτερμαιερ είναι ο πρώτος από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγητές για τη συνεργασία. Είχαμε πολύ καλές συναντήσεις οδών πριν από τα Χριστούγεννα και δώσαμε πολλά στοιχεία για την ενδιάμεση έκθεση. Σας ευχαριστώ που τα λάβατε υπόψη. Θα ήθελα να τονίσουμε τρεις τομείς όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε μερικές αλλαγές. Στο 1.3 Μιλάμε για τις ε, βασικές ε, νομικές διευθετήσεις όπου τα χρήματα εξαφανίζονται από το σύστημα και νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο των καταπιστευμάτων, διότι δεν διέπονται από καμία διαφάνεια και χρησιμοποιούν άλλα μέσα που δεν είναι ανοιχνεύσιμα σε σχέση με τους φορείς. Μιλάμε για τις τράπεζες και τους ρυθμιστές, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για τους ε, νομικούς συμβούλους και για αρχές που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις. Ξέρετε ότι στο Γιβραλτάρ υπάρχει μια ειδική δραστηριότητα η οποία δεν είναι ανιχνεύσιμη όπως αναφέρεται και σε ένα βιβλίο το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε αυτές τις δραστηριότητες και στο 2,1 στη νομική κατάσταση, στο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά πόσο θα πρέπει να επεκταθούμε κάπως και επίσης ως προς τις δικαιοδοσίες οι οποίες δεν συνεργάζονται. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Ένα από τα πρώτα ζητήματα όταν αρχίσαμε με τις εργασίες μας αφορούσε την ΦΑΤΚΑ, τον είπα. Ακούσαμε τι υπόθηκε στην ακρόαση και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο συστήματα όπως το ΦΑΤΚΑ είναι πραγματικά αποτελεσματικά. Προσβλέπω στη συνεργασία μας Νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες μάθαμε πολλά και κατά τις αποστολές θα μάθουμε πολύ περισσότερα. Ελπίζω να με υποστηρίξετε, να μας υποστηρίξετε. Ευχαριστούμε τον κύριο Λινίντερ Μάιο. Έχουμε τον κατάλογο των σκιωδών. Ο κύριος Άγγελ Τσαμπάτσκι τώρα με βάζει αυτόν τον κατάλογο. Αλλά δεν είναι παρόν. Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Φάβιο Ντιμάζη. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ τον σκιώδη μας που θα έλεγα ότι είναι 50% έγκυος και δεν μπορεί να παρευρεθεί. Ευχαριστώ τους συζητητές για την ε, πολύ καλή εργασία τους. Θα εστιάσω κυρίως ε, στα σημεία όπου θέλει να εκφράσει κριτική η ομάδα μου, αλλά να μην δώσω τη λάθος εντύπωση. Πολλά σημεία μας βρίσκουν σύμφωνος, αλλά προτιμώ να εστιάσω στα σημεία που θεωρώ ότι ακόμη υπάρχουν κενά. Ένα μεγάλο έλλειμμα στην εργασία μας είναι κάτι για το οποίο δεν φταίει κανείς μας. Είναι κυρίως αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητήσαμε πρόσβαση σε κάποια έγγραφα και δεν μας έχει ακόμη παρασχεθεί. Ενώ ήδη λειτουργούμε για αρκετό χρονικό διάστημα. Και αυτό οπωσδήποτε έχει επιπτώσεις και για την εργασία μας ε, επί της εκθέσεως. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό. Πρώτα απ' όλα για τις διαστάσεις του σκανδάλου του, των εγγράφων του Παναμά νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούν πιο συγκεκριμένα μερικές ε, εγκληματικές δραστηριότητες όπως ε, η παράνομη διακίνηση ατόμων και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για να καταστεί σαφές ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Για το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, δηλαδή στο κεφάλαιο 2, θα θέλαμε να αναφερθούμε για κάποιες ε, μεταφορές πόρων που αποφεύγει, όπου αποφεύγεται εντελώς η φορολόγηση. Δηλαδή κάποιοι πόροι φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχουν φορολογηθεί και μετά καταλήγουν σε φορολογικούς παραδείσους. Δεν είναι δηλαδή θέμα μόνο αναπτυσσόμενων χωρών και εμείς πρέπει να κάνουμε την εργασία που μας αναλογεί. Τώρα για το νομικό πλαίσιο όσον αφορά τους ενδιαμέσους. Πρέπει να θέσουμε το θέμα των κυρώσεων Ξέρουμε ότι παίζουν ε, χρήσιμο ρόλο οι ενδιάμεσοι αυτοί. Πολλοί ακόμη συμμετέχουν ε, στην ε, σύνταξη της νομοθεσίας για αυτά τα περίεργα νησιά. Γιατί δεν έχουν οι δήμονες τα νησιά αυτά για να εκπονήσουν νόμους. Οι ενδιάμεσοι λοιπόν θα πρέπει και αυτοί να υπόκεινται σε κυρώσεις δεν πρέπει να υπολοιπόμεθα αυτών που υπόθηκαν στην Επιτροπή Τάξε. Γιατί και εκεί διατυπώθηκαν συστάσεις για αυτά τα θέματα. Για το κεφάλαιο 3, η μεταφορά του νομικού πλαισίου στην εθνική νομοθεσία. Ωραία, σωστό, αλλά να, να δούμε και το γεγονός ότι οι φορείς επιβολής του νόμου, οι εφορίες και τα λοιπά Πολλές φορές δεν έχουν επαρκές ε, προσωπικό. Επίσης και ε, όσον αφορά την επιβολή της ποινική νομοθεσίας υπάρχουν κενά. Πρέπει να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Στο κεφάλαιο 4, η διεθνής διάσταση, πολύ καλό θα ήταν να αναφερθούμε και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Γιατί προφανώς ε, είναι από τους πιο βασικούς ε, παράγοντες. Τώρα έχουμε ένα πρόεδρο που θέλει να κάνει την Αμερική και πάλι μεγάλη χώρα, αλλά δεν συμμορφούνται με τις αρχές της αμοιβαιότητας, δηλαδή δεν εφαρμόζουν ε, τις κοινέ προδιαγραφές για την υποβολή εκθέσεων. Και τώρα για τις κυρώσεις να πούμε ότι μπορούν να υπάρχουν, θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες εκκυρώσεις και αντίμετρα για τις χώρες που δεν συνεργάζονται. Νομίζω στο προηγούμενο έγγραφο εργασίας υπήρχαν τέτοιες αναφορές που τώρα δεν περιλαμβάνονται. Ήδη ψηφίσαμε για τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση Επιτροπής γιατί δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη. Οπότε Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις εταιρείε και άλλες δομές ε, που έχουν οικονομική δραστηριότητα από αυτές τις δικαιοδοσίες. Θα τους επιτρέπουμε να έχουν δοσοληψίες και οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Και τέλος, πρέπει να δούμε το θέμα των αρμοδιοτήτων των εξεταστικών επιτροπών. Ξέρουμε τα όρια μας. Πιστεύω ότι είναι καλό να ε, έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την ΑΦΚΟ. Και αυτό θα βοηθήσει τους συναδέλφους μας σε άλλες εξεταστικές επιτροπές στο μέλλον. Γιατί είμαι σίγουρος ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν σκάνδαλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να επιτρέψουμε στο Κοινοβούλιο να τα αντιμετωπίσει καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. ο συνάδελφος Βαγκίγκολ από τους Πράσινους. Προοδευτική οικονομική επιστήμη έχει διάφορες, ε, διάφορους κλάδους. Ε. Αυτό που είπε ο Φάμπιο για το 50% έγκυος δεν το έχω ξανακούσει πρέπει να σας πω. Ε, θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι εννοείτε αγαπητέ συνάδελφοι. Εγώ πάντα νόμιζα ότι είναι κανείς έγκυος ή όχι. Τέλος πάντων, όσον αφορά το έργο μας, πιστεύω ότι το έγγραφο εργασίας αντικατοπτρίζει ε, αυτά που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Αν το συγκρίνετε δε με την εντολή της Εξεταστικής Επιτροπής, μπορέσαμε ε, μέχρι στιγμής δυστυχώς να διερευνήσουμε λίγα πράγματα γιατί η βασική εντολή μας είναι να εξετάσουμε αν τα ευρωπαϊκά όργανα όχι ε, η φορολογική παράδειση ή κάποια ενδιάμεση τα, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα και αν τα κράτη-μέλη ε, τήρησαν τις σχετικές υποχρεώσεις τους. Και αν υπήρξαν περιπτώσεις κακοδιοίκησης. Ε, μέχρι στιγμής ε, το έγγραφο αυτό έχει τη μορφή ενός εγγράφου πολιτικής ε, στο οποίο θα καταλήγουμε σε συγκεκριμένες συστάσεις. Δεν θέλω να προκαταβάλω την συζήτηση. Αυτά που είπατε σε κάθε περίπτωση είναι σωστά. Εμείς δεν διαφωνούμε. Αυτό που μας ανησυχεί όμως είναι ότι έχουμε μια εντολή η οποία παραθέτει τομείς ενδεχόμενης κακοδιοίκησης και ενδεχόμενων νομικών παραβιάσεων. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να συνδέσουμε την εντολή μας με τα ευρήματα των εργασιών μας. Και αυτό δεν ε, μέχρι στιγμής επαρκώς στο έγγραφο εργασίας. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ε, εξετάσουμε και να λάβουμε υπόψη μας τις νομικές μας υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένης και τις υποχρεώσεις συνεργασίας που κατοχυρώνεται στη συνθήκη και στη συνέχεια να ε, προχωρήσουμε στο ουσιαστικό έργο ε, της αξιολόγησης των, ε, ε, των ε, διερευνητικών εργασιών που έχουμε κάνει και στη συνέχεια να συγκρίνουμε τα ευρήματα αυτά με εκείνα που προέκυψαν από ακροάσεις, από έγγραφα κτλ. κτλ. Ωστόσο, δυστυχώς η DG Just δεν μας έχει στείλει τίποτα, μας έχει στείλει άσχετα έγγραφα, η Tax δεν μας έχει στείλει τίποτα Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το Συμβούλιο μάλιστα έχει συμφωνήσει να μην συνεργαστεί αποτελεσματικά με εμάς. Νομίζω αυτό είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Σικλούνα, με τον οποίο συζητήσαμε χθες, φαίνεται ότι είναι ε, συνεπή η στάση του Συμβουλίου να μην συνεργάζεται μαζί μας και γι' αυτό και δεν ήρθε σήμερα εδώ προφανώς προκειμένου να μην υποβληθεί σε εξέταση από εμάς. Αυτό είναι το βασικό ε, αντικείμενο της, δικές, της δικής μας Επιτροπής. Να βρούμε τα έγγραφα προκειμένου να μπορέσουμε να, να αποδείξουμε ότι πράγματι υπήρξαν περιπτώσεις κακοδιοίκησης και παραβιάσεις της νομοθεσίας. Και καθώς λοιπόν δεν έχουμε στη διάθεσή μας τα έγγραφα που χρειαζόμαστε, χρειάζεται να βασιζόμαστε περισσότερο στις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τους συνεισηγητές και τη γραμματεία να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο τις, ε, τα δημοσιεύματα του ICIJ στα μέσα ενημέρωσης, ακριβώς γιατί εκείνοι έχουν πρόσβαση στα ε, αυθεντικά έγγραφα που εμείς δεν έχουμε. Δυστυχώς το ICIJ δεν μας έδωσε τα έγγραφα στα οποία έχουν εκείνη πρόσβαση παρότι τα είχαμε ζητήσει, παρόλα αυτά έχουν προβεί σε δημοσιεύματα σε πάνω από 80 χώρες. Αδύνατον να κάτσουμε εμείς ως ευρωβουλευτές να τα διαβάσουμε όλα, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση και μια αξιοποίηση των όλων ε, ευρημάτων των, ε, της Διεθνούς Σύμπραξης ε, Ερευνητών Δημοσιογράφων. Αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα ε, και πολιτικής φύσης όπως ε, ανακοίνωσες και εσύ χθες ή προχθές. Ε, ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Και πιστεύω ότι πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση. Είναι επίσημη απόφαση να λάβουμε τα έγγραφα αυτά, αλλά υπάρχουν τρία κράτη-μέλη ε, που μας έχουν ε, υποσχεθεί ότι ε, θα μας αποστείλουν έγγραφα. Δεν είναι μεταξύ αυτών όμως εκείνες οι χώρες που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Άρα και, μάλλον και θα χρειαστεί να, να την θητεία μας. τα, ονόματα αν μας τα δίνατε ενδεχομένως να μπορούσατε να, να ασκήσετε μια μεγαλύτερη πίεση. Όχι δεν έχω ακριβή κατάλογο αυτή τη στιγμή Ξέρω ότι η Γαλλία και η Γερμανία και οι κάτω χώρες ε, είναι πρόθυμες να μας ε, παράσχουν έγγραφα, ε, οι άλλες όχι. Μπορεί όμως κάτι στο μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα δηλαδή να έχει αλλάξει. Βουλγαρία και Σλοβακία επίσης μαθαίνω, μάλιστα. Ωραία. Η FDD δεν εκπροσωπείται, η NF, η κυρία Κάπελ επίσης δεν είναι εδώ. Catch the eye διαδικασία. Όποιο θέλει μπορεί να πάρει τον λόγο. Ο Λουί Μισελ έχει ήδη ζητήσει τον λόγο. Κάριος Ροζάτη στη συνέχεια. Und Catalan Ivan. Bitte. <coughs> Monsieur le Président, cher. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι συμμερίζομαι τις απογοητεύσεις του προλαλήσαντα σε σχέση με τα μέσα που διαθέτουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην εντολή μας. Είμαι πολύ ανησυχός γιατί αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι με τα έγγραφα που λείπουν, δηλαδή έλλειψη πληροφόρησης ε, για να θέσουμε τα πραγματικά ερωτήματα που μας απασχολούν, θα αντιμετωπίσουμε παράλληλα και ένα θέμα μεθοδολογίας. Δεν οφείλεται σε εσά, κύριε Πρόεδρε, εσείς προσπαθείτε να εργαστείτε σωστά, αλλά στην ε, προηγούμενη συνεδρίαση μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αφήνουμε τους παρεμβαίνοντες να ξεφύγουν από τις απαντήσεις. Εγώ δεν έλαβα απαντήσεις. Η μόνη απάντηση που έλαβα ήταν ότι από τη δική τους πλευρά όλα βαίνουν καλώς το σύστημά τους είναι ασφαλές, έχουν εσωτερικούς ελέγχους για να μπορέσουν να ελέγξουν την προέλευση του χρήματος. Αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε, να απαντήσουμε. Δηλαδή δεν θα έχουμε τις σωστές ε, συστάσεις τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν απαρεγκλήτως οι κυβερνήσεις. Δηλαδή υπάρχει πολλή δεοντολογία, αλλά πολύ λίγες συστάσεις εν της πράγμαση. Αναρωτιέμαι κατά πόσο δεν θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των προσκεκλημένων, έτσι ώστε να μπαίνουμε στην ουσία και να μπορέσουμε να τους κολλήσουμε στον τοίχο. ο, όταν ο κύριος Μανάρ, Μανάρτ νομίζω, μίλησε, εκπροσωπεί τους νομικούς συμβούλους και τους δικηγόρους. Όταν μας λέει ότι δεν είναι εμπλεκόμενοι, αυτό με σοκάρει. Δηλαδή πρόκειται για ψέμα, κατάφορο ψέμα, κάτι το οποίο δεν μπορώ να δεχτώ. Αναρωτιέμαι κατά πόσο μεταξύ μας δεν θα πρέπει να έχουμε μία προσυνεννόηση για να ξέρουμε ποιος θα υποβάλει ποιο ερώτημα για να μπούμε στις λεπτομέρειες, για να είμαστε μία πραγματική εξεταστική ε, επιτροπή. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο πέρα. Πρέπει να πιέσουμε τους ανθρώπους να απαντήσουν, τους εμπλεκόμενους, τους προσκαλεσμένους. Οι συγητές κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, ειλικρινά, δεν θα καταλήξουμε κάπου. Οι δύο παρεμβαίνοντες ε, ήταν ο Πάλαν και η κυρία Άλλινγκτον ήταν πολύ, παρουσίασαν πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Έδειξαν ότι θέλουν να μας βοηθήσουν. Πράγματι, είναι αξιόπιστοι. Θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους σε βάθος. Ως προς τις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει μια εξαιρετική έκθεση της ε, υψηλής ομάδας για τις παράνομες ροές χρημάτων από την Αφρική. Ο Τόμας Μπέκι, ο πρώην πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής, ήταν ο πρόεδρος και νομίζω ότι θα πρέπει να τον καλέσουμε για να μας επεξηγήσει το όλο θέμα. Γιατί τον είχαμε καλέσει στο παρελθόν, τον πρώην πρόεδρο Μπέκη και πραγματικά η έκθεση αυτή είναι αρκετά καλογραμμένη και τεκμηριωμένη. Θα ήθελα να την κοινοποιήσετε στα μέλη. Υπάρχει στα εγγραφά μας είναι, πρόσφατη, είναι πρόσφατο αυτό το έγγραφο και πραγματικά θα μπορούσε να μας εμπνεύσει για την περαιτέρω εργασία μας. Επίσης για τη ΦΑΤΚΑ θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να καλέσουμε ενδιαφερόμενος. Ως προς το καθεστώς μας, το δικό μας καθεστώς λειτουργίας, θα πρέπει να βασιστούμε σε συγκεκριμένες συστάσεις. Ζήτησα συγκριτικούς πίνακες για την νομοθεσία στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν έχω λάβει ακόμα αυτούς τους πίνακες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα δούμε που υπάρχουν οι ελλείψεις και ποιες είναι οι χώρες που δεν τηρούν τους κανόνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μισελ. Καταλαβαίνω α, ότι ορισμένοι είπαν ότι όλοι οι ομιλητές ε, προχθές ήταν καλοί. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν όλοι καλοί όμως. Ο πρώτος ε, γύρος ε, των ομιλητών ήταν καλός, αλλά στο δεύτερο γύρο μόνο ο εκπρόσωπος της Price Waterhouse Cooper είχε ένα καλό επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας. ή άλλοι απλώς απέφευγαν τις ερωτήσεις, αλλά δεν έχουμε καμία δυνατότητα να τους υποχρεώσουμε. Και φυσικά, αν μας στείλετε το έγγραφο για την Αφρική, θα το δούμε. Και ίσως θα μπορούσατε να ασκήσετε την επιρροή σας για να βελτιωθεί η συνεργασία μας με την ε, βελική κυβέρνηση. Ήσασταν πρώην εξωτερικό. Να Είναι λοιπόν η έκκληση που κάνω προς εσάς προσωπικά. Η διαδικασία είχε συμφωνηθεί με τους συντονιστές και τη τηρήσαμε. Είπαμε ότι αν υπάρξουν ε, μεμονωμένες περιπτώσεις θα επιχειρήσουμε να καλέσουμε και άτομα που ίσως θα ήσαν διατεθειμένα να μας πούν κάτι και όχι απλώς να αποφεύγουν τις ερωτήσεις. Συμφωνώ όμως ότι την Τρίτη αυτό συνέβη. Αλλά το θέμα είναι λοιπόν να έχουμε διαμορφώσει τις ερωτήσεις ε, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα όταν κάποιος ε, συζητάει μια συγκεκριμένη υπόθεση να μπορεί να ε, την διερευνήσει σε βάθος. Μέχρι στιγμής ε, δεν το επιτύχαμε. Είμαι ωστόσο πολύ ευχαριστημένος με την εργασία των δύο συνσηγητών, γιατί είναι παρόντες, γιατί κάνουν καλές προτάσεις και γιατί έτσι βελτιώνουμε το σύστημα. Ο επόμενος στο κατάλογό μου είναι ο Ντάριος Ροζάτη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ε, συνεισηγητές μας που προετοίμασαν αυτό το έγγραφο. Είναι μια θαυμάσια αφετηρία. Η μόνη γενική παρατηρήση που έχω να κάνω είναι ότι ίσως να είναι υπερβολικά φιλόδοξο. Καλύπτει πολλούς τομείς, πολλά θέματα. κατά τη γνώμη μου θα είναι ε, μάλλον δύσκολο να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά, δεν θα, υπάρχουν, δεν θα υπάρξει επαρκής χρόνος. Και ίσως ε, να μην υπάρχει και αρκετός χρόνος για όλα αυτά. Καλύτερα λοιπόν να εστιάσουμε στα πιο σημαντικά θέματα, τα πιο κρίσιμα της εντολής μας. Να κάνω μια σύντομη απαρίθμηση των καθηκόντων που προτείνουν φιλόδοξα οι συνεισηγητές μας για το τελικό κείμενο της έκθεσης. Η επίπτωση των επιπτώσεων στα, στους ε, προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Αρνητικές επιπτώσεις στα, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Να εξετάσουμε τις στατιστικές ε, ισοζυγίου πληρωμών για να δούμε αν υπάρχουν ύποπτες ροές πόρων κατάλογος ε, χωρών υψηλού κινδύνου και τα κριτήρια με τα οποία θα ορίζεται ο υψηλός κίνδυνος. Μία επισκόπηση της νομοθεσίας ε, που υπάρχει για τη φοροδιαφυγή και του νομικού πλαισίου στα κράτη-μέλη. εξετάσουμε συγκεκριμένες υποθέσεις, να μελετήσουμε υποθέσεις να εξετάσουμε τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών. Αδυναμίες ε, του νομικού πλαισίου στις αναπτυσσόμενες χώρες που οδηγούν σε αυτές τις ε, ροές κεφαλαίων. Οι κανόνες μας για αυτούς που καταγγέλουν παρανομίες. Όλα αυτά πολύ σημαντικά θέματα. Αλλά δεν ε, είμαι σίγουρος ότι θα προλάβουμε να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά τα θέματα και να καταλήξουμε σε αποτελεσματικές συστάσεις. Πιστεύω θα έπρεπε να περιορίσουμε περισσότερο το φάσμα των θεμάτων που θέλουμε να δούμε. Ορισμένες ερωτήσεις έχουν απαντηθεί αλλού από τον ΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη ή από αυτό το FATF αυτό είναι το πρώτο μου γενικό σχόλιο. Κατόπιν. Να ξαναδούμε πώς ε, διαρθρώνεται αυτό το κείμενο. Θα ενεθάρρυνα τους συνεισηγητές να εξετάσουν μια κάπως διαφορετική δομή. Θα μπορούσαμε να διαιρέσουμε το κείμενο και άρα και την έκθεση σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο θα περιγράψει γενικά το φαινόμενο φοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής μέσω φορολογικών παραδείσων και μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών. Το πρώτο τμήμα λοιπόν θα δώσει στατιστικά στοιχεία να ορίσει το μέγεθος του προβλήματος και τη ζημία στους εθνικούς προϋπολογισμούς και κάποιες άλλες επιπτώσεις αυτών των κακών πρακτικών. Δεύτερο, να περιγράψει τους μηχανισμούς, τις δομές τις συνήθεις συμπεριφορές για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς γίνονται στην πραγματικότητα αυτά τα πράγματα. Τρίτο κομμάτι θα έπρεπε να εξηγήσει τα αίτια που προκαλούν αυτά τα παραθυράκια, αυτές τις αδυναμίες, να αποτιμήσουμε το νομικό πλαίσιο και να εντοπίσουμε τις κύριες αδυναμίες του, υπαρχον, του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, γιατί το κύριο πρόβλημα είναι αυτή η υπερβολική μυστικότητα που επιτρέπεται από το νομικό πλαίσιο ορισμένων χωρών και επειδή δεν εφαρμόζεται σωστά ο νόμος ή επειδή απλώς παραβιάζεται. Τρίτο αυτό λοιπόν, δηλαδή να εντοπίσουμε τα αίτια και νομικά και οικονομικά και όλους τους παράγοντες που διευκολύνουν ε, την, ε, το ξέπλυμα του χρήματος, τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή. Και τέταρτο φυσικά οι συστάσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα του ενωσιακού δικαίου, στις εθνικές νομοθεσίες, τα προβλήματα που έχουμε κατά τη μεταφορά του ενωσιακού νόμου στις εθνικές νομοθεσίες, τι μπορούμε να κάνουμε παγκόσμια, διεθνώς, και βεβαίως και τις ενδεχόμενες κυρώσεις κατά των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών. Νομίζω ότι μια τέτοια δομή, τέσσερα τμήματα, θα μας επέτρεπε να εστιάσουμε στα σημεία που είναι ζωτική σημασίας για την εργασία μας. Ευχαριστώ. Να προσθέσω και ένα πέμπτο κεφάλαιο. Πρόταση για την ε, ε, μετεξέλιξη του δικαίου για την διερεύνηση. Να έχουμε δηλαδή την δυνατότητα να καλούμε ε, υποχρεωτικά δηλαδή ε, ανθρώπους εδώ και να μην ε, εξαρτώμαστε από την ε, καλή τους βούληση. Ε, εδώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταρτήσουμε και μια σύσταση για το πώς θα μπορούσε να μεταξελιχθεί τέλος πάντων το ισχύον δίκαιο. Ράμον Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες υποδείξεις ε, για αυτό που θα ήθελα να περιληφθεί σε αυτή την έκθεση. Χαίρομαι για το προσχέδιο και σας ευχαριστώ για την εργασία σας, για την εργασία των συγητών. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι ως προς τις συστάσεις, όχι ως προς την περιγραφή του φαινομένου, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες εγγράφων και βιβλίων που περιγράφουν τι συμβαίνει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως όπως είπε και ο εισηγητής, θα πρέπει να ορίσει έναν οδικό χάρτη για το τι υποδεικνύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διεθνή κοινότητα και αρχές. Ως προς τις υποδείξεις συστάσεις, θα ήθελα να προσθεθεί μία, δηλαδή οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι διάφοροι ενδιάμεσοι που αποτιμούν την κατάσταση να πρέπει να μην εργάζονται σε αυτή την μεσολάβηση με τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε για να μπορέσουμε να ανασχέσουμε κάπως αυτές τις οντότητες, αυτούς τους οργανισμούς. Γιατί είναι ένα θέμα κοινωνικής ευθύνης. Επίσης η Ευρώπη θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή την φορολόγηση συναλλαγών, διότι Όσο περισσότερη ρύθμιση υπάρχει, τόσο και μεγαλύτερη διαφάνεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Επίσης, λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια μιας εντολής που αντιβαίνει την αποδοτικότητα. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί, αλλά στον τομέα της φορολόγησης Δυστυχώς τα κρατη φέρουν την ευθύνη και λειτουργεί το Συμβούλιο με ομοφωνία. Άρα όλες μας οι συστάσεις προσκρούν σε μία οντότητα που είναι το Συμβούλιο. Υπάρχει ένας περιορισμός επίσης της ομοφωνίας στη φορολογική πολιτική και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει εναρμόνιση και αποδοτική πολιτική κατά της φοροδιαφύγης τη στιγμή που έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη. Από το 2014 το Κοινοβούλιο έχει προβάλει μία πρόταση ρύθμισης των εξεταστικών επιτροπών. Εγώ είμαι εισηγητής στην Επιτροπή συνταγματικών υποθέσεων και δυστυχώς οι εξεταστικές μας επιτροπές δεν έχουν αποκλειστικές αρμοδιότητες διότι προσκρούμε πάντα στο Συμβούλιο. Άλλοι τρεις ομιλητές, πρωτού ξαναδώσουμε το λόγο στους δύο συνεισηγητές, Καταλήν Ιβαν, Έλλη Σλάιν και μετά Σαν Γκίγκολτ. Παρακαλώ. Ιβαν. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ότι θα πρέπει να τονίσουμε τρία ζητήματα που είναι ύψης της σημασίας. Καταρχήν, θα πρέπει να αξιολογήσουμε το νομικό πλαίσιο που διαθέτουμε, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε νομοθετικά και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μόνο τότε θα δούμε κατά πόσο χρειαζόμαστε περαιτέρω νομοθέτηση ή προσαρμογή της νομοθεσίας. Μέχρι τότε προβάλλουμε ιδέες, αλλά δεν συμβαίνει και τίποτα έμπρακτα. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την, τον πολυσχηδή χαρακτήρα των, δραστηρι... των υπεράκτιων δραστηριοτήτων, όπως και των ενδιάμεσων υπάρχουν συμβουλευτικές εταιρείες σε διάφορα επίπεδα. Μπορούμε να έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση, μια μεγάλη εταιρεία. Σε δεύτερο επίπεδο υπάρχουν ε, χιλιάδες και σε τρίτο επίπεδο υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις ε, συμβουλευτικής. Και γι' αυτό ακριβώς αυτές οι επιχειρήσεις αποκόπτονται από την μητρική και λένε και έτσι η μητρική μπορεί να πει «Α, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτές τις ε, υπεράκτιες δραστηριότητες». Επίσης, το τρίτο ζήτημα αφορά τις υπηρεσίες ε, πληροφοριών και πάταξης του οικονομικού εγκλήματος. Υπάρχουν ε, αυτές οι υπηρεσίες σε αρκετές χώρες, σχεδόν σε όλες, αλλά δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πάταξης του οικονομικού εγκλήματος στα 28 κράτη-μέλη, 27 στο εγγύς μέλλον. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία εργασία συντονισμού στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ε, καλέσαμε αυτή την ε, υπηρεσία του Λίχτενστάιν μέσα στα πλαίσια μιας ακρόασης και είχα την εντύπωση ότι δεν υπάρχει και διάθεση συντονισμού αυτών των δραστηριοτήτων και των ε, υπηρεσιών πάταξης οικονομικού εγκλήματος. Δεν υπήρχε τέτοια διάθεση επί της ουσίας. Η Egmont Group, που ε, πολλές φορές βρίσκονται και συναντώνται αυτές οι υπηρεσίες δεν θέλει να συμμετάσχει. Και πέρα από την Egmont Group κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ιδίω η συνεργασία με την Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού ε, τις, ε, τις ε, διατάξεις για τις μονοπρόσωπες εταιρείε, όλα αυτά είναι πολύ ζητήματα, αλλά ο κύριος Κοσάτη είπε δικαίω ότι είναι τόσο ευρύ το πεδίο της υπόθεσης που δεν μπορεί χρονικά αλλά και απόψη περιεχομένου μια εξεταστική επιτροπή να τα καλύψει όλα. Το γνωρίζαμε αυτό εξ αρχής, το γνωρίζαν και οι συνεισηγητές. Μπορώ να πω κάτι για μια παρέμβαση του καθηγητή Πάλαν που είπε χθε ότι περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε, ε, σε παράγωγα ε, κρύφτηκαν σε τέτοιου είδους εταιρείε. Η ονομαστική αξία ε, αυτών των ε, παραγωγών ε, ανέρχεται σε 683 εκατομμύρια δολάρια. Ε, βλέπετε ότι προφανώς τα δεδομένα και τα μεγέθη είναι τεράστια και υπερβαίνουν και τις ε, ε, δυνατότητες της δικής μας Εξεταστικής Επιτροπής. Γι' αυτό και χρειάζεται συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων. Κυρία Σλάιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές που κατάρτισαν ένα πολύ καλό κείμενο, καλή βάση εργασίας το οποίο μου φαίνεται πλήρες. Βεβαίως θα πρέπει να εμβαθύνουμε ορισμένα επιμέρους σημεία και χαίρομαι γιατί λαμβάνουμε υπόψη την παγκόσμια διάσταση του ζήτηματος. Ο Λουί Μισελ το προανέφερε όταν προανέφερε το έγγραφο της Αφρικανικής Ένωσης που παρουσιάστηκε από τον πρώην πρόεδρο Μπέκη στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Θα πρέπει να δούμε τι μας λένε τα έγγραφα. Τι μας δείχνουν τα έγγραφα του Παναμά. Μας δείχνουν πώς με ένα απλό κλικ τάχιστα μεταφέρονται τεράστια ποσά από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Και ένα άλλο ουσιώδες ζήτημα. Εμείς φυσικά έχουμε μία ελιπέστατη εντολή. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε. Αυτό είναι άκρος απογοητευτικό. Γιατί τη στιγμή που το θέμα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, το οποίο είναι παγκόσμιο, γιατί αφορά την ε, μεταφορά αυτών των κεφαλαίων και το γεγονός ότι μπορεί κανείς να επιλέξει την δικαιοδοσία που του προσφέρει συνθήκες απορρίτου, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ορίων μας. Τη στιγμή όμως που δεν έχουμε τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που θα θέλαμε, ακόμα και για την πρόσβαση στα έγγραφα, θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας και να δείξουμε και εφευρετικότητα για παράδειγμα, η πρόταση της Επιτροπής για το Country by Country Reporting, εάν μας δίνει στοιχεία όχι σε επίπεδο συνόλων σε, ευρωπαϊκή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν μας δίνει λοιπόν στοιχεία ως προς τις επιχειρήσεις που δρούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαμε να επεκταθούμε. Ο Σβέν και ο Φάμπιο μιλούσε για εγκυμοσύνη κατά 50%. Αστιεύτηκαν επ' αυτού. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να βασιστούμε σε αυτό τον κατακαιρματισμό της πληροφορίας για να έχουμε μία πληροφόρηση έστω και κατά 50%. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είμαι αισιόδοξη γιατί ως προζητήματα ζωτικής σημασίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πέρσι το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα επ' αυτού, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα αν δεν υπάρχει μία διεκυβερνητική δομή σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε και οι αναπτυσσόμενες χώρες να πρέπει να ε, λαμβάνουν το λόγο και να συμμετέχουν ισότιμα σε σχέση με την αναθεώρηση των φορολογικών κανόνων. Έτσι θα έχουμε μία πλαισίωση έτσι ώστε κανένας, καμία από αυτές τις χώρες να μην είναι εκτεθειμένη. Ευχαριστώ κύριε Σλάιν. Έχετε δίκιο όσον αφορά το διεθνές πλαίσιο. Ο κύριος Ντεμάζη το ανέφερε ήδη ότι γίνονται μεταφορές πόρων ε, που δεν φορολογούνται και παίζει ρόλο, συμμετέχει δηλαδή και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ρόλο και το γεγονό ότι ζητήθηκε από την Apple στην Ιρλανδία να πληρώσει 13 δι συμπληρωματικό φόρο, αυτό οφείλεται όμως και ε, σε ένα παραθυράκι του Αμερικανικού νόμου που επιτρέπει κάπου να βάλει κανεί ε, ε, σε ορισμένους φορολογικούς παραδείσους κάποιους πόρους οι οποίοι φορολογούνται μόνο όταν επανέλθουν. Είχαν παρκάρει έτσι 30 δις και το η Apple στην ουσία εκβίασε την Αμερικανική κυβέρνηση και τους είπε «Κοιτάξτε, 38% δεν πληρώνουμε, αλλά αν χαμηλώσετε το συντελεστή θα επανέλθουν οι πόροι αυτοί». Αυτά τα χρήματα όμως συνολικά είναι 130 δις, αν ο νέος Αμερικανός πρόεδρος αποκαλύψει αυτή τη δυνατότητα και μειώσει το συντελεστή για να επανέλθουν αυτοί οι πόροι, τότε στην ουσία κλείνουμε ένα πολύ σημαντικό παραθυράκι. Και γι' αυτό το ζητάμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αντιμετωπίσουν αυτά τα παραθυράκια που βεβαίως ε, καθίστανται δυνατά μόνο λόγω και ευρωπαϊκών ε, κενών στην νομοθεσία. Ο κύριος Γκίγκολτ. Κοιτάξτε, το βασικό θέμα είναι τι θέλουν οι πολίτες να ψάξουμε εμείς να βρούμε. Βεβαίως ε, πρέπει να έχουμε ευρύ πνεύμα Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι θα βρούμε ψάχνοντας. Γι' αυτό ήθελα να είναι ευρεία η εντολή. Αλλά ποτέ δεν είχα την πρόθεση ούτε την ε, ψευδέστηση ότι θα μπορούσαμε να τα καλύψουμε όλα. Πρέπει όμως να έχουμε ευρεία προσέγγιση. Ανοιχτό πνεύμα. Αλλά ποιο είναι το βασικό στοιχείο της εντολής μας. Γιατί υπάρχει ένα παράλληλο σύστημα που οι απλοί πολίτες θα το θεωρούσαν περίεργο. Σωστά υπόθηκε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτός ο παράλληλος μυστικός κόσμος που σίγουρα αντιβαίνει το πνεύμα του νόμου και ορισμένες φορές συχνά θα έλεγα και κατά του γράμματος της ε, νομοθεσίας κατά της ε, λεύκανσης χρήματος του ξεπλήματος χρήματος και καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής ε, δραστηριότητας στον πλανήτη. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν δράσει αποτελεσματικά για να σταματήσει αυτό το παράλληλο σύστημα. Που σημαίνει ότι για πολλούς δεν ισχύει το κράτος δικαίου. Η εντολή μας λοιπόν είναι ποιος έχει και ποια κράτη-μέλη συγκεκριμένα έχουν εμποδίσει την εφαρμογή του νόμου. την ε, ουσιαστική επιτήρηση της εφαρμογής του νόμου δηλαδή. Γιατί δεν συνέβη αυτό. Γιατί δεν άλλαξε η νομοθεσία, γιατί δεν προτάθηκαν αλλαγές στην νομοθεσία, ούτω ώστε η πράξη να συμβαδίζει με το πνεύμα της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης ε, παρανόμων πόρων. Αυτό το θέμα τέθηκε από τα έγγραφα του Παναμά. Και αυτό είναι το ερώτημα. Ποια κράτη-μέλη δεν εφάρμοσαν στην ουσία τον νόμο και γιατί δεν τόλμησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους κυνηγήσει. Ε, έχουμε ακούσει διάφορες προφάσεις. Ότι ορισμένοι ενδιαφέρονται μόνο για το γράμμα του νόμου. Μεταφέρονται οι οδηγίες, αλλά μετά δεν ελέγχουμε εάν στην πραγματικότητα Και αυτή την εργασία πρέπει να την κάνει το FATF και άλλοι οργανισμοί και χαίρομαι πως Νάλφο Ήβαν τόνισε ότι ούτε αυτοί οι οργανισμοί στην ουσία κάνουν σωστή δουλειά. Και κάποιοι εκεί, κάποιοι ελάχιστοι καημένοι στην Κομισιόν, στην DigiJust, έπρεπε να εξετάσουν ε, πώς λειτουργεί το 5% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Αυτό πρέπει να θέσουμε. Γιατί δεν έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση τα τελευταία 20 χρόνια. Ευχαριστώ. Ε, σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα παίζει και η ομάδα εργασίας για τον κώδικα διοντολογίας, το έργο της οποίας μπλοκαρίστηκε τα τελευταία χρόνια πολλές φορές από διάφορα κράτη-μέλη. Θέλω να αναλάβω μια πρόταση από το πάνελ 1. Ένας ομιλητής λοιπόν είπε ότι οι δικηγόροι, οι διάμεσοι, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παραβιάζουν το πνεύμα του νόμου χωρίς να παραβιάζουν το γράμμα του. Και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά μια διαπίστωση κλειδί για το πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αλλαγές. Πρέπει να οξύνουμε την, ε, ομοθεσία, προκειμένου ακόμη και η καταστρατήγηση του πνεύματος του νόμου να διώκεται. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο, οπότε δίνω το λόγο στου δύο συνεισηγητέ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ ε, ε, συνάδελφοι. Νομίζω ότι πραγματικά είχαμε μια πολύ γόνιμη ε, συζήτηση σήμερα που αποδεικνύει επίσης ότι η εντολή μας φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων είναι ευρεία ε, και αυτό βεβαίως ε, ε, καταδεικνύει την ανάγκη να εργαστούμε παρά την έλλειψη πρόσβασής μας σε όλα τα έγγραφα. Εμείς λοιπόν εργαστήκαμε παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Και αυτό είναι και το δίλημα, ξέρετε, ότι στην πραγματικότητα το καλύτερο θα ήταν να έχουμε πρόσβαση στα πραγματικά έγγραφα, στα αυθεντικά έγγραφα, για να δούμε που, σε ποιες περιπτώσεις ε, τα κράτη-μέλη και τα όργανα δεν κατάφεραν να ε, εφαρμόσουν την νομοθεσία και στη συνέχεια να καταλήξουμε σε συστάσεις. Πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο εκ παραλλήλου, γιατί ακριβώς δεν έχουμε πρόσβαση ακόμη. Και γι' αυτό έχει και αυτή τη μορφή το έγγραφο εργασία μας. Συμφωνώ πάντως με το γεγονός ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην εντολή μας, την κακοδιοίκηση, εφαρμογή της νομοθεσίας και παραβιάσεις αυτού και να δούμε ε, με ποιους τρόπους υπήρξαν πραγματικά στοιχεία που χρειάζεται να αναφερθούν στην, ε, ε, στην τελική μας έκθεση. Ο κ. Νίτερμαϊερ είπε θέλουμε να εξετάσουμε και εμείς αυτή την ιδέα της, ευρωπαϊκή, της ευρωπαϊκής φάτκα. Ε, χρειάζεται να κάνουμε και επιτόπιες επισκέψεις θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα εκεί που θα πάμε και η δική μου προσέγγιση είναι να είμαστε ανοιχτοί και να κάνουμε μια συλλογική δουλειά όλες οι πολιτικές ομάδες, να εξετάσουμε όλες τις προτάσεις και να ε, καταφέρουμε να καταλήξουμε στις πιο αποτελεσματικές, τις οποίες και θα εντάξουμε στο έγγραφο εργασίας. Ομάδα για τον κώδικα διοντολογίας το είπατε κι εσείς, και στην τάξη 1 και στην τάξη 2 καλέσαμε να γίνει μια ε, γενική μεταρρύθμιση του κώδικα διοντολογίας για την φορολογία των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταργηθεί το, η αρχή του απορρίτου, της ανωνυμίας, που είναι μεγάλα προβλήματα, γιατί ξέρουμε ότι ε, αυτό μας έχει εμποδίσει να καταπολεμήσουμε ε, επιζήμια καθεστώτα φορολογικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ολόκληρη η, δομή της ε, ομάδας αυτής για τον κώδικα διοντολογίας μας εμποδίζει εμάς τους ίδιους να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τα ζητήματα της φοροποφυγής και φοροδιαφυγής στην ενιαία αγορά. Μετά, το είπε ο Φάβιο Μάτση νομίζω, για την ε, παρακράτηση φόρου. Το είχαμε αναφέρει και στις δύο εξεταστικές επιτροπές τάξη 1 και 2. Χρειάζεται να δούμε ποιε συστάσεις έχουμε ήδη καταρτήσει και έχουν υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο στις άλλες δύο εξωτερικές ε, και, και τι έχουν κάνει ε, αντιστοίχως οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Ποιε συστάσεις μας δηλαδή έχουν ήδη υιοθετηθεί. Ε, δεν συμφωνώ με το να κάνει το, συμβούλιο, το κοινοβούλιο συστάσει και στη συνέχεια αυτές να τις αγνοούν εκείνοι που πρέπει να τι εφαρμόσουν. Και μια τελική παρατήρηση σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή. Είχαμε μια συνάντηση και με τον Αμερικανό εκπρόσωπο της Γερουσίας και συζητήσαμε το πώς εκείνοι ε, διοργανώνουν αυτές τις εξετατικές επιτροπές. Ε, μας ενέπνευσε, ε, μας ενέπνευσαν τα όσα μας είπαν και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε και σε συστάσεις για το πώς θα μπορούσαν να συγκροτούνται στο μέλλον τέτοιου είδους εξεταστικές επιτροπές με αποτελεσματικότερο τρόπο ε, να εξασφαλίζεται βεβαίω η πρόσβαση στα έγγραφα και φυσικά υπάρχει και το ε, ζήτημα της, ε, του, του δικαιώματος κλήτευσης και του δικαιώματος εξέτασης του Κοινοβουλίου, που πράγματι υπάρχει πρόβλημα ε, όσον αφορά τη συνεργασία μας και με τα κράτη-μέλη και με το Συμβούλιο. Αυτά, να δώσω το λόγο και στον συνάδελφο Πέτερ και στη συνέχεια, τέλος να πω βεβαίως ότι θα λάβουμε υπόψη μας ε, στο έργο μας όλα τα σχόλια που έγιναν. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και οικοδομητική η συζήτηση και με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πίτερ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Θα ήθελα να σταθώ σε μερικές από αυτές για να φτάσουμε σε πιο γενικά συμπεράσματα. Ο κύριος Μάιερ, είπε για τους μεσάζοντες και μίλησε για τους δικηγόρους περισσότερο. Άλλοι είπαν ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις τράπεζες, ενώ άλλοι μίλησαν για τους φορολογικούς συμβούλους και τις φορολογικές εταιρείες, λογιστικές εταιρείες. Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο έδαφος και μετά να κάνουμε μια βαθύτερη έρευνα ανάλογα με τις έρευνες. Αν δούμε ότι οι ενδιάμεσοι μεσάζοντες θα πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο, θα πρέπει να το κάνουμε ανάλογα με τα ευρήματά μας. Εάν άλλα ζητήματα είναι πιο περιθωριακά, θα τα αφήσουμε στην άκρη. Και το ίδιο ισχύει και για αυτά που είπε ο Φάμπιο Ντεμάση που μίλησε για διεύρυνση του πλαισίου του εγγράφου, ο κύριος Ροζάτη ζήτησε συρρήκνωση. Άλλοι θέλουν περισσότερη, άλλοι λιγότερη φιλοδοξία. θα πρέπει να αρχίσουμε με ένα ευρύ πλαίσιο το οποίο σιγά σιγά θα περιορίσουμε. Ακόμα και οι Μάση και Ντεροζάτη έχουν δίκιο όταν αναφέρουν ότι το κείμενο αυτό θα μπορούσε να διευρυνθεί, θα μπορούσε να δούμε και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τα τέσσερα σημεία που προανέφερε ο κ. Ρωσάτη υπάρχουν στο έγγραφο. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτο και κάπως γενικευμένο και ανάλογα με τα ευρήματά μας θα εστιάσουμε την προσοχή μας εκεί που πρέπει. Ο Σβέν είπε ότι αυτό το έγγραφο θα μπορούσε να συζητηθεί και σε επίπεδο συντονιστών. Πολλές φορές ε, λείπουν έγγραφα και από τα κράτη-μέλη και αν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για έλλειψη συνεργασίας, για μη διάθεση συνεργασίας, θα μπορούσαμε σε μια συνέντευξη τύπου ε, και στο Συμβούλιο να ζητήσουμε αλλαγή αυτής της τάσης να συμμετέχει περισσότερο ο τύπος, η ΜΚΟ, για να κάνουν τη ζωή δύσκολη στους πολιτικούς που δεν συμμορφώνονται. Αλλά καταρχήν θα πρέπει να δούμε τα αποδεικτικά στοιχεία ως προς την έλλειψη συνεργασίας εκεί που υπάρχει. Αυτά έχω να πω και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν τελειώσαμε ακόμα εντελώς γιατί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε η κυρία Μαρίνα Βάιταους η οποία εργάζεται για φορολογικά θέματα στη Γενική Διεύθυνση του κυρίου Μοσκοβισή. Εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Φορολόγησης για το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας. Να σας ενημερώσω για την κατάσταση των εγγράφων γιατί φαίνεται πολύ σημαντικό από ό,τι φαίνεται και για την Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω ότι τα έγγραφα τάξη 1 και 2 θα χορηγηθούν τις επόμενες μέρες στην Επιτροπή σας. Ε, να σας εξηγήσω γιατί η διαδικασία πήρε τόσο χρόνο. Τα έγγραφα αυτά τα είχαμε δώσει στην τάξη 1 και τάξη 2 ε, με, με διαφορετική νομική βάση και επειδή η ΠΑΝΑ συστάθηκε με βάση την απόφαση του 1995 χρειάστηκε να υπάρξει και πάλι διαβούλευση των κρατών μελών για τα ίδια έγγραφα και η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε πέρυσι το Δεκέμβριο. Μια άλλη προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να χορηγήσει εμπιστευτικά έγγραφα στην Επιτροπή σας ήταν ότι έπρεπε να υπογραφεί ο διακανονισμός που προτείναμε που ήταν ταυτόσιμος με το διακανονισμό για την έμις και την τελική μορφή του υπογεγραμμένου γράφου τη λάβαμε πολύ πρόσφατα γιατί υπήρξαν κάποιες περιτέρω, περαιτέρω ε, αιτήσει από κάποια μέλη να δοθούν και στους ε, διαπιστευμένους βοηθούς τα έγγραφα αυτά. Έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, τα αντιμετωπίσαμε και η Επιτροπή σας δέχτηκε το διακανονισμό στις 30 Ιανουαρίου, λέει η ομιλήτρια. Α, στις 13 εννοεί. Και από ό,τι φαίνεται όλες οι υπηρεσίες της Επιτροπής ε, αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν την αποστολή αυτών των εγγράφων και υπενθυμίζω ότι με βάση την απόφαση του 1995 τα έγγραφα εφόσον προέρχονται από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σταλούν μετά από διαβούλευση και πάλι με τα κράτη-μέλη, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από την Επιτροπή η αποστολή αυτών των εγγράφων. Ελπίζω οι εξηγήσει αυτές να διευκρινίζουν την ε, υποεξέλιξη αυτή η διαδικασία και όπως σας είπα η Επιτροπή έχει κάθε διάθεση να συνεργαστεί με την Επιτροπή σας και η εργασία είναι σε εξέλιξη στις υπηρεσίες της Κομισιόν για να ε, ε ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Ευχαριστώ κυρία Βάιταους από άποψη χρόνου ε, και χρονοδιαγράμματος ε, έχουμε φτάσει στο σημείο που πραγματικά χρειαζόμαστε πλέον τα έγγραφα. Έχουμε υποβάλει τα αιτήματά μας εδώ και εβδομάδες, μήνες. Υπήρξαν πράγματι κάποια προβλήματα, αλλά πλέον είναι πραγματικά καιρό, ε, το έχουμε συζητήσει και με τη Γραμματεία. Ε, στην επόμενη συνεδρίαση Ολομέλειας ε, στο Στρασβούργο θα συζητήσουμε στις 13 Φεβρουαρίου θα, θα συζητήσουμε με τους συντονιστές τι ε, μέτρα ε, θα ήταν αναγκαία αν δεν έχουμε ακόμη μέχρι εκείνη τη στιγμή τα έγγραφα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συζήτηση, για τη συνεργασία, ευχαριστώ τους συνεισηγητές, ε, όλους τους συναδέλφους που ήταν εδώ. Κυρίσω την λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Επόμενη συνεδρίαση είναι σήμερα το απόγευμα στο, στην αίθουσα ε, ένα G3, 2 με 4 ε, ε, το απόγευμα, το workshop με ευθύνη διοργάνωσης του κυρίου Κόφοντ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους Δερμήνη.